η ψηφοφορία θα έπρεπε να επαναληφθεί για το λόγο αυτό. Ευχαριστώ. Yeah, Κύριε Γκόλνης, το θέμα αυτό το συζητήσαμε. Το επαληθεύσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή με βάση τον κορονισμό η απόρριψη του κυρίου Σιμανσκή, τον κύριο από τον κύριο Σιμάνσκι ήταν γνωστή στους περισσότερους. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν ε, είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε η εκθέση του Σιμάνσκι. Και όπως και να έχει, Έχουμε ένα άρθρο 171 παράγραφος 5 το οποίο μιλάει ξεκάθαρα και λέει ότι όταν, ότι ο πρόεδρος, ο προεδρεύων της προφορίας κρίνει την εγκυρότητα της ε, ψηφοφορίας και αυτή η απόφαση είναι ανέκλητη. Κυρία Αποδηματά προείδρευε, αποφάσισε ότι ανέγκυρη ψηφοφορία δεν γίνεται τίποτε περαιτέρω. Δεν υπάρχει δυνατότητα να προσβληθεί αυτή η απόφαση. Κυρίε και κύριοι, θα είδατε ίσω σήμερα μία προβολή στο, στην είσοδο του Λούις Βάις με εικόνες για την αποφυλάκηση των δημοσιογράφων που κρατούνται στη Συρία. Με, αυτό, με αυτή την εκδήλωση θέλει το Συμβούλιο να αποστείλει ένα μήνυμα προς τους δημοσιογράφους αυτούς και τις οικογένειές τους, δεν τους έχουμε λησμονήσει και τους υποστηρίζουμε με κάθε δύναμη. Η Συρία είναι σήμερα μάλλον ε, κατά πάσα πιθανότητα ο πιο επικίνδυνος τόπος για δημοσιογράφους. Έχουν ε, χάσει τη ζωή τους ε, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πάνω από 100. Είναι κρατούμενοι πολλοί, σε ομοιρία, έχουν πολλοί εξαφανιστεί και μένουν αγνοούμενοι για μήνες πολλοί πολίτες από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, συμπολίτες μας δηλαδή. Και νομίζω ότι όπως και εγώ όλοι σας θαυμάζετε το θάρρος που δείχνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να μας προσφέρουν πληροφόρηση, για να εξυπηρετήσω αυτό το δικαίωμά μας στην πληροφόρηση. Τρία χρόνια ένας φρικτός εμφύλιος πόλεμος με κλιμάκωση της βιαιότητας, για τον οποίο δεν θα είχαμε καμία ενημέρωση χωρίς την αυτοθυσία αυτών των δημοσιογράφων. Θα ξέραμε τίποτα για τους ε, πολέμους, για τις βιοπραγίες, για τις φαγές, ε, για την βία που ασκείται βάρος των παιδιών, για όλα τα προβλήματα και τα δεινά που αντιμετωπίζει ο λαός της Συρίας. Ανεξαρτήτως λοιπόν του αν κάποιος προέρχεται από την ε, Ευρώπη ή τη Συρία ή από οπουδήποτε αλλού, αυτοί οι δημοσιογράφοι που κρατούνται πρέπει να απελευθερωθούν, να αποφυλακιστούν. Το απαιτούμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Έκθεση της κυρίας η κυρία Φερέρα είναι ασθενής. Σήμερα εκπροσωπείται από τον κύριο Σάνσες Πρεσέντο. Της ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Και δίνω το λόγο στην κυρία Μπόλτσο, πρόεδρο της Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να εξηγήσω γιατί ζητάμε αναβολή του νομοθετικού ψηφίσματος, ούτω ώστε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, με την